Okay. Dear colleagues, please take your seats. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. Okay, dear colleagues, please take your seats. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Now, uh, where's the no. Uh, as uh, as uh, some of you know. Όπως ίσως γνωρίζετε ορισμένοι από εσάς, όπως ίσως γνωρίζετε κάποιοι από εσάς. Πριν από τέσσερις ημέρες ορίστηκα νέος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ. Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης αυτής ήταν ότι την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, όταν για πρώτη φορά επισήμω συνείδησα του ομολόγου μου από τι χώρε σας, κανεί δεν με συνεχάρει. Όλοι μου είπαν «Καλή σου τύχη». Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω μόνο ένα σύντομο αντίο. Θα μου λείψει πάρα πολύ το κοινοβούλιο. Όλοι οι φίλοι που έκανα εδώ θα μου λείψουν πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο μέρος στην Ευρώπη γιατί το κοινοβούλιο συνδυάζει και πάθος και συμπόνια και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και δεν θέλω να είναι στα αγγλικά το τελευταίο αντίο. Και επειδή δεν θέλω να ξεχάσετε τα ελληνικά που μάθατε το τελευταίο 1,5 χρόνο, θα σας προτείνω να κάνουμε το εξής. Πώς είναι το υπέρ στα ελληνικά? Υπέρ. How do we say against? Against. Κατά. Κατά. How do we say abstention? Αποχή. Very good. Okay, now, hold a second, Mr. President. What I want is... Ωραία. Λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα. Οι σοσιαλιστές και εγκούε υπέρ. PPE, κατά. Ε, εσείς το ΕΛΚ και η Συντηρητική πάντα κατά. Η πράσινη και η φιλελεύθερη αποχή. Απλό, ωραία, πάμε. Let's go. Fantastic. Fantastic. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σούλτ ζητάει το λόγο για διαδικαστικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Απορρίπτεται, λέει ο κύριο Σούλτ στα ελληνικά. Ε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ ε, να μου δώσετε το λόγο, διότι σίγουρα έχω την κατανόηση των συναδέλφων, ε, μιλώντας εξ ονόματο της ομάδας μας, αλλά νομίζω και όλων των συναδέλφων, να σας πω ότι εσείς Κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνετε ένα βαρύ φορτίο, το γνωρίζετε καλύτερα από εμά έχετε την πλήρη αλληλεγγύη μας για τα νέα σας καθήκοντα, γιατί όλοι μας, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας θέσεις, έχουμε όλοι μια επιθυμία και ευχή αυτή η θαυμάσια χώρα της οποίας είστε υπουργό εξωτερικών το συντομότερο και ή δυνατό με τη βοήθειά μας να ξεπεράσει τη βαθιά της κρίση. Τη χρειαζόμαστε την Ελλάδα, είμαστε αλληλέγγυοι και με εσά και με τη χώρα σας και θα ήθελα προσωπικά να σας πω κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών και αγαπητέ Σταύρο ότι ήσασταν και είστε όχι μόνο φίλος αλλά καταπληκτικός συνάδελφος πάντα για μας πλούτος σας ευχαριστώ πολύ για τα τόσα χρόνια συνεργασίας και καλή σου τύχη Σταύρο Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι χαίρετε και τώρα το λόγο έχει η ε, ε, Αξιοθαύμαστε Αντιπρόεδρος, κυρία Νταγιάννα Γουάλης. Ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία.